Liebe Kolleginnen und wir sollten Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολύ φιλόδοξες λίστες ψηφοφορίας. Οι ε, συνάδελφοι, ή ε, ε, μάλλον η συνάδελφος έρχεται, της οποίας την έκθεση θα ψηφίσουμε. Ελπίζω μέχρι να έρθει η ώρα να την ψηφίσουμε να έχει έρθει. Ε, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη καταρχάς έτσι όπως είναι. Υπάρχουν αντιρρήσει, θέλετε να την αλλάξουμε, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι από ό,τι βλέπω, οπότε εγκρίνεται. Σημείο 2. Έγκριση των, ε, ε, πρακτικών της Επιτροπής ε, της 10ης Οκτωβρίου. Βρίσκεται στους φακέλους σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Άρα προτείνω ω συνήθω να θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά εγκρίνονται σε περίπτωση που μέχρι το τέλο τη σημερινή συνεδρίαση δεν έχουν υπάρξει αντιρρήσει. Πάμε στο 3. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Έχουμε διερμηνία στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, τσεχικά, εστονικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Και να σας θυμίσω βεβαίως ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Πάμε στις ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε δύο εκθέσεις, δύο γνωμοδοτήσεις και ξεκινούμε με την έκθεση πρωτοβουλίας, εκπαίδευση στην ε, ψηφιακή εποχή, προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για, την, ε, για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η συγγήτρια η Γιάννα Τόμ. Γιάννα, θέλεις μήπως το λόγο? Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ένα ευχαριστώ μόνο για όλους. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Άρα πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία και ξεκινούμε με τη συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 13 προς 11, εγκρίνεται. 92, υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ, πιο καθαρά τα χέρια σας να τα βλέπω. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, καλύτερα έτσι. 93, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται να το εξετάσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 138. Πέρας ψηφοφορίας. 16 προς 9. Εγκρίνεται. 193. 139, ε, συγγνώμη. Α, συμβαστική 13. Διορθώνει η πρόεδρος. Συμβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 133. αρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 13-12. Απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, είναι λίγο τεμπέληδες οι σοσιαλιστές σήμερα, μου φαίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 156. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 176. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 181 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 182 υπέρ. Α, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 181. Πέρας ψηφοφορία. 17 προς 8. Εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το δούμε ηλεκτρονικά και αυτό. Ψηφίζουμε την 183. Πέρας ψηφοφορίας. 14 προς 8. Εγκρίνεται με 5 αποχές. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. 8. λάθο. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά αποχές νομίζω να το δούμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 58 ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας 16 προς 11 εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Λάθος. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην ε, Ήτρε. Όχι, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε αυτή. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 26 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται ομόφωνα συγχαρητήρια Γιάννα. Και ευχαριστώ εσένα και τους σκιώδεις εισηγητές σου για τη δουλειά που κάνατε. Πάμε στην επόμενη έκθεση. Das ist der Entwurf... Σχέδιο Έκθεση για το νέο θεματολόγιο για τον πολιτισμό. Η ο κύριος Γραμματικάκης. Θέλετε το λόγο? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τη συνεργάτη μου τη Χριστίνα Μερκουριάδη αλλά και όλους τους συναδέλφους γιατί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την έκθεση και είχαμε 180 τροπολογίες. Νομίζω ότι με πολύ κόπο και πολύ καλή συνεννόηση πετύχαμε να φτάσουμε σε ένα αξιόλογο τελικό σχέδιο και για πρώτη φορά αν ψηφιστεί σήμερα θα έχουμε μια, ένα δρόμο προς τον πολιτισμό της Ευρώπης που ελπίζω κυρία Πρόεδρε και με τις δικές σας προσπάθειες να γίνει λεωφόρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία λοιπόν. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40, 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 και 64 ταυτόσημες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 73, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90, 90 και 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 94 υπέρ, όχι, 93, την 94 την ψηφίζουμε, 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το δούμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 16 προς 11 εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 και 155 Ταυτόσιμες. υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνονται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές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 Okay, also an Stelle habe ich einen Fehler. Κάπου έκανα λάθος. Στην 85, ε, στη σελίδα 5, ε, ε, εγκρίθηκε, αλλά ψηφίσαμε και την 86, την οποία δεν έπρεπε να έχουμε ψηφίσει. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά, 2 εποχές. Με μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν ε, εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Bericht. Das ist der Entwurf einer Stellungnahme. Πάμε στην ε, επόμενη έκθεση. Ε, σχέδιο για την ε, διαβίβαση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Ο κύριος Ζωγοράκης είναι ο εισηγητής. Συνάδελφε, θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Δεν έχω να πω κάτι. Να συνεχίσουμε στις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Wunderbar. Τέλεια. Προχωράμε λοιπόν αμέσως. Πάμε στην τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ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 αποχές, απορρίπτονται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά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 Την 13, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 14 προς 11, απορρίπτεται. 113, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114 και 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 121 και 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 123 και 124 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 125 και 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Την 127. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18-8. Εγκρίνεται. Δεν το είχα καταλάβει, συγγνώμη. 15 ε, και 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά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 αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές. Να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τρία άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Όχι, τώρα πέρα ψηφοφορία. 12 προς 15 απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές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 αποχές απορρίπτεται, 64 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 65 και 66 είναι ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται, 67 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 68 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 69 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 70 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 και 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 και 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. 24 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφο κατά και τρεις αποχές. Ομόφωνα εγκρίνεται η εκθεσή σας. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Μάλιασε η γλώσσα μου. Πάμε στο σχέδιο ε, γνωμοδότησης για την εκπόνηση του προγράμματος InvestEU. Εισηγητής ο συνάδελφο Τζαμπάσκι. Είναι εδώ, όχι, θέλετε το λόγο. Πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ 73 να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 73. Geschlossen. Πέρασε ο Συγγνώμη. 14 προς 12 απερίφθη. Πάμε στην 74. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 80 υπέρ. Κατά. Θα, ψηφί... θα καταψηφίσεις την ε, τροπολογία σου. Είμαστε στην 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά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 Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την συμβαστική 5 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία, ναι όντω. είχατε δίκιο. 10 προ 17 απορρίπτεται και ζητώ συγγνώμη. Προχωρούμε. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται 96 συνάδελφοι να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 23 προς 3 εγκρίνεται Πάμε στην 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 100 και 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές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 αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 23 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε στην 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την συμβαστική πρόταση 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 15 προς 11 εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 Αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική 9, υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. 41, υπέρ, κατά, αποχές, δεν κατάλαβα, νομίζω εγκρίνεται, αλλά στα αριστερά μου δεν είδα πολλά χέρια. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 41 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφορίας ε, εντάξει, 27, 0. Ευχαριστώ. Ε, τι, καμιά φορά. Μάλλον ε, κουράστηκα. 40, όχι, συμβαστική 10, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 47, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει, βλέπω πολλά κόκκινα φωτάκια. Μάλλον πέρας ψηφοφορίας. Ναι, 21-5. Απερίφθη. 51 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Αυτή πάλι δεν κατάλαβα αν εγκρίνεται ή όχι. Πάμε να τη δούμε ηλεκτρονικά. Αρχίτη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 51. Πέρας. 14 προς 13 απορρίπτεται. Ε, εντάξει, δεν ήταν ε, εύκολο να το καταλάβω. Πάμε στην 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. και πέρας. 25 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή εγκρίνεται με τεράστια πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τα καταφέραμε. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν τόσο συγκεντρωμένοι. Und wir machen auch sofort weiter. Και συνεχίζουμε αμέσω Και πάμε στο σημείο 10 τη σημερινή διάταξη. εξέταση της, του σχεδίου έκθεσης για την ε, δημιουργία του προγράμματο Creative Europe. Η συγκίτρια, η συνάδελφο Σίλβια Κώστα. Ε, ε, προθεσμία για την, ε, για την υποβολή τροπολογιών 29 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτισμού στις 20 Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς. Σίλβια, σου δίνω το λόγο να μας παρουσιάσεις την έκθεση. Έχεις 5 λεπτά. Θα επιχειρήσω, Πρόεδρε, να μείνω εντός των 5 λεπτών να ευχαριστήσω θερμά για την υποστήριξη, για τη συνεργασία, την πολύ καλή συνεργασία με τους κοιόδης. Ε, συναντηθήκαμε με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς. Ε, να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής, αλλά και την Κομισιόν, τη ΓΑΜΑ η οποία ήταν απολύτως διαθέσιμη και έτοιμη να μας βοηθήσει. Τώρα, να θυμίσω κάποια σημαντικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα αυτό που είναι το μόνο άμεσο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολιτιστικά και οπτικοστικά θέματα. Διατήρησε λοιπόν την αυτονομία του και τη δομή του, τις στοχεύσεις του επίσης και δεν ενσωματώθηκε ή διαλύθηκε όπως και άλλα ε, εντό άλλων προγραμμάτων και άλλων πλαισίων. Αυτό το υπογράμμισαν και οι ενδιαφερόμενοι φορέ. Ε, περισσότερο για τα θέματα πολιτισμού παρά για θέματα οπτικοακουστικά και μέσων. Αυτό το είχαμε πει και στην ενδιάμεση έκθεση και την έκθεση αξιολόγηση ε, ε, θεωρώ πάντως ότι το συνολικό πλαίσιο πηγαίνει προς τη θετική κατεύθυνση αλλά δεν είναι επαρκώς λεπτομερές και πολλέ από τις ε, τροπολογίες τις δικές μας, άνω των 100 εξάλλου, ε, είναι στοχευμένε προ την κατεύθυνση αυτή ε, και βάσει των συνομιλιών που είχαμε με όλους του ενδιαφερόμενου. Τώρα, η φιλοδοξία του προγράμματο αυτού που είναι πολύ ευρύτερη από εκείνου του προεπταετία, εάν δεν βασίζεται σε σε χρηματοδοτικού πόρου, θα είναι απογοητευτική η αποτελεσματικότητα. Ε, και επομένω και στην ενδιάμεση έκθεση ε, και στο ψήφισμα για το ΠΔΠ του περασμένου Μαρτίου ως Κοινοβούλιο ε, είχαμε ζητήσει αυτά που ζητώ και ως εισηγήτρια τα 2,8 δισεκατομμύρια και όχι τα ονομαστικά που αναφέρει η Κομισιόν ή στην πρότασή της. Και θεωρώ και ελπίζω ότι σε αυτό θα έχουμε τη δέσμευση και του, του ολόκληρου του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τώρα, για τα διατομεακά, για την παιδεία, για τον πολιτισμό δεν πρέπει να μιλούμε για συνολικά μεγέθη, αλλά ποσοστία 33, ε, 25 αν όξαμε καλά και τα λοιπά για τα υπόλοιπα των τομέων. Τώρα, αυτό το της συνεργασίας που είναι το πιο σημαντικό για τους κοινωνικούς φορείς και τους ενδιαφερόμενους πρέπει να είναι τουλάχιστον 70% ε, για να εξασφαλίζεται και ένα επαρκές επίπεδο επιτυχίας. Για, γενι... για τους γενικούς στόχους πέραν το 2, κοινωνικό και οικονομικό, έχω προσθέσει και την αναγνώριση της ε, εγγενούς αξίας του πολιτισμού, δηλαδή τις ειδικότητες που εμπίπτουν στον ειδικό αυτό κλάδο τομέα, εκτός των καλλιτεχνών. Ε, δεύτερον, επανεισήγαμε την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία ω προπόθεση ε, στήριξη του προγράμματο που δεν υπήρχε περιέργω, αλλά και από τη βάση των ε, εμπειριών που είχαμε τον τελευταίο χρόνο, είχαμε συζητήσει και νωρίτερα, υπογραμμίζοντας και την ε, συμμετοχικότητα, την έννοια, την αίσθηση τη συμμετοχικότητας για του πολίτε και για το αφήγημα το ευρωπαϊκό που είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τους πολίτε. Τώρα, για τους στόχους ε, συμφωνούμε με την Κομισιόν για το Seal of Excellence, αλλά θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο, λίγο πιο απτό. Δηλαδή, για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις αρχές διαχείρισης, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις στοχεύσεις, τα έργα δηλαδή εντός του προγράμματος που, ε, που εμπίπτουν στη χρήση της φραγίδας αυτής ποιότητας, ώστε να αναγνωρίζεται. Τώρα, πολιτισμός και μέσα επικοινωνίας. Συμφωνούμε με τις οριζόντιες και τομεακές δράσεις, είναι πιο διαθρωμένες από την νωρίτερα, είναι σημαντικά αυτά. Έχουν εισακουστεί κάποιες από τις προτάσεις μας για ειδική προ... πίστοση, τέλος πάντων πρόβλεψη για την μουσική, κάποια ε, καινοτόμα έργα στο πλαίσιο των ε, πολιτισμικών, ε, μεγαλύτερη προσοχή στην αξιοποίηση των εκδόσεων και όχι μόνο των μεταφράσεων και προβλέπουμε τρία κριτήρια για τις ενισχύσεις υψηλή πολιτιστική αξία, αντίκτυπος και ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή. Τα εφαρμοστικά έργα ε, μάλλον τα έργα συνεργασία. Ε, θέτουμε, ε, την, ε, υπογραμμίζουμε τη σημασία της τοπικής αξίας και προσθέτουμε και τα μικροέργα και θεωρούμε ότι πρέπει να επανέλθει και η βράβευση, μάλλον η ενίσχυση για το Ευρωπαϊκό Θέατρο που δεν υπάρχει πια. Μέσα τώρα. Είναι, δεν είναι εξέλιξη, αυτό είναι υπό εξέταση, αλλά εν πάση το τα οπτικοακουστικά εγώ εισήγαγα ε, μία παραπομπή ε, στα κινηματογραφικά, στα ντοκιμαντέρ, ε, στα θεατρικά, ε, εισήγαμε την, ε, έννοια των φίλων, όπως και στα προϊόντα και μέσα της τηλεόρασης. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τους παραγωγούς και διανομής, τους ανεξάρτητους για να αποφύγουμε και ε, τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ συγκεκριμένων υποκειμένων. Τώρα, το διατομιακό πλέον συμβαίνει αυτό, γίνεται σιγά σιγά αυτό που θα έπρεπε να είναι, δηλαδή πολλαπλών ειδικοτήτων και με μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα του πλουραλισμού και θα λέγαμε έτσι της δημοσιογραφίας ποιότητος. Και να κλείσω με μια νέα αναφορά στο θέμα, στη διεθνή διάσταση μάλλον, γιατί εγώ προτείνω να το πούμε Creative Europe Mundus για τις δράσεις που έχουν ε, ε, μια διάσταση διεθνή, αν θέλετε, και τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που θα πρέπει κανείς να δει σε ένα παρατηρητήριο που θα είναι αφιερωμένο στα θέματα του πολιτισμού. Μέχρι στιγμής έχουμε δει πολύ λίγα στην ε, κατάσταση αυτή. Και τέλο, στο Invest Youth InvestEU, you, με συγχωρείτε, λέει ο μιλήτρια τελικώς, ε, συνενώνει 15 διαφορετικά μέσα. Εδώ έχουμε προσθέσει όμως κάποιες ανησυχίες που είχαν ανακύψει, δηλαδή στον κανονισμό θα πρέπει να ε, ε, εισαχθούν όλες οι προτεραιότητες, όλα τα κριτήρια και όλες οι συνθήκες εκείνες και προϋποθέσεις που είχαμε εγγυηθεί στους διάφορους φορείς των ε, ε, ε, της παραγωγής των οπτικοακουστικών μέσης, θεωρούμε ότι ε, η Econ, η Invest EU και τα λοιπά θα πρέπει να εμπίπτουν στους τομεακούς κανονισμούς σχετικά με τις στοχεύσεις και τα κριτήρια για να μην χάσουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα που είχαμε επιτύχει ε, προηγουμένως. Θα μείνω εδώ και περιμένω περαιτέρω ε, παρατηρήσεις από τους συνάδελφους. Ευχαριστώ Σιλβία. Πάμε στους χειώδες συγκητές τώρα. Ξεκινούμε με το ΕΛΚ. Η Ζαμπίνα νομίζω θα αναλάβει. Ε, εντάξει δεν θα την αναλάβω ακριβώς, θα εκπροσωπήσω τον συνάδελφο. Θα παρουσιάσω αυτά που έκανα από τη δική του την πλευρά και θα διαβάσω τα τελευταία του λόγια εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί ε, πλέον ε, θα είναι δήμαρχος στην πόλη του οπότε είναι τα τελευταία του λόγια εδώ. Καταρχά να ευχαριστήσω την κυρία Κώστα για το σχέδιο έκθεσή τη και για τη δουλειά που έκανε για αυτό το σημαντικό πρόγραμμα. Το πιο σημαντικό βεβαίω σημείο είναι ο διπλασιασμό του προπολογισμού του, του τρέχοντος προγράμματος Creative Europe και το καλωσορίζουμε. Συμφωνώ επίσης για τις περισσότερες ε, λεπτομέρειες που πρέπει να υπάρξουν για την εφαρμογή, για την συμπληρωματικότητα για τι συνέργειε μεταξύ των ε, προγραμμάτων χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως την ε, σφραγίδα Αριστεία και το Invest EU. Μία από τι βασικότερε προκλήσει τη τρέχουσα ε, πρόταση είναι να εγγυηθούμε την διευκόλυνση για του πολιτιστικού και του τομεί δημιουργία. Η εγγύηση αυτή έχει περάσει στον κανονισμό InvestEU πια. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν οριζόντιε αναφορέ με τον κανονισμό InvestEU και αυτές να προσθεθούν στο κείμενο. Συμφωνώ με την νέα δομή για, τον, για την πτυχή της, ε, του πολιτισμού που θα εισαγάγει οριζόντιους και, τομεακούς, ε, οριζόντιους και τομεακές δράσεις, κυρίως ό,τι αφορά την, τις νέες οριζόντιες δράσεις για την χρήση της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του κλάδου. Ένας από ε, Ήμουν ένας από τους ε, συγγραφείς του ε, συγκεκριμένου νομικού πλαισίου, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε έτσι την πρόταση ε, Creative Europe και τη σχετική έκθεση. Ε, έτσι θα μπορέσουμε να ε, συμπληρώσουμε την ε, πρόταση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία με ανησυχούν. Το ΕΛΚ πάντα ήταν ιδιαίτερο υποστηρικτικό για τους τομείς της δημιουργίας και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση του κυρίου Μόργανο και στην έκθεση του κυρίου Έλερ και βεβαίω υποστηρίζουμε την ιδέα να ενισχύσουμε τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων δημιουργικών οργανισμών και των χαρασόντων την πολιτική για να ενισχύσουμε τον διάλογο με του εκπροσώπους του κλάδου. Στο νέο σχέδιο έκθεση προτείνουμε να υπάρξει ένα παρατηρητήριο για τον τομέα των δημιουργικών τεχνών, αλλά φοβούμαι ότι αυτό θα σήμαινε μεγάλο κόστο δεδομένου το ότι ο προπολογισμό μα είναι ήδη πολύ περιορισμένο. Και για μένα οι λεπτομέρειε ε, για τη δομή και για τη χρηματοδότηση αυτής της, ε, αυτού του φορέα δεν είναι σαφεί. Νομίζω ότι μπορούμε να ε, εμπιστευτούμε την αποστολή αυτή σε υπάρχοντε οργανισμού. σω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μα δώσει μια ιδέα για το πώ θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη εμπειρογνωμοσύνη για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τον αντίκτυπο των πολιτικών πολιτισμού και να έχουμε καλύτερα ποσοτικά οικονομικά και πολιτικά αποτελέσματα. Το άλλο σημαντικό σημείο είναι η δομή του προγράμματο. Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε στην πρόταση τη Κομισιόν και να διατηρήσουμε τη γενική δομή του τρέχοντο προγράμματο με, τις, με τους τρεις πυλώνες, πολιτισμός, ΜΜΕ και διατομεακά θέματα. Και αυτό λαμβάνει υπόψη και τις, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τι συγκεκριμένες ανάγκε των διαφόρων τομέων και ακολουθεί τι θετικέ εξε, εξελίξεις που είχαμε στα πλαίσια του τρέχοντο προγράμματο. Με την ε, τροπολογία 34 για, την, για, την, ε, για τον πολιτισμό περιλαμβάνουμε και, περιλαμβάνουμε και τα οπτικοακουστικά project, αλλά για σκοπούς δημοσιονομικούς και διοικητικούς, δεδομένου του ότι θα είχαμε δύο διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει που ασχολούνται με το ίδιο φάκελο, μπορεί τα πράγματα να είναι λίγο περίπλοκα. Τέλο, για τα μικρά project, έχω κάποιε αμφιβολίε για την τροπολογία 61 και την οικονομική συμβολή του προγράμματο που θα πρέπει να φτάνει στο ανώτερο το 80% του κόστου τη επιχείρηση, όπω γράφεται στην ε, πρόταση ε, και ο διαγωνισμό θα πρέπει να δώσει μικρά project με υψηλότερο βαθμό χρηματοδότηση από σε μεγάλα project. Ε, εμείς γενικώ θέλουμε να έχουμε πολλά μικρά project, αλλά μας ενσυχεί λίγα και αυτή η αναφορά, γιατί θα πρέπει να έχουμε ισορροπία, αλλά και να διασφαλίσουμε την ευελιξία και την ποιότητα για όλα τα σχέδια. Το ΕΛΚ θα προετοιμάσει τροπολογίες και θέλουμε φυσικά ε, να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την ε, κυρία Κώστα και τους υπόλοιπους σκιώδες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Σαμπίνε. Ο κύριος Διάκονο έχει το λόγο. Παρακαλώ. Τρία λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι προθέσεις είναι καλές, αξιέπαινο αυτό. Έχουμε συνεργαστεί πολύ θετικά με την κυρία Κώστα μέχρι τώρα και ελπίζω θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχω μια πρόταση, μια σύσταση για τη σημερινή συζήτηση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Μιλάμε για επενδύσεις στον τομέα της, του πολιτισμού. Οι επενδύσεις μεταφράζονται σε νούμερα. Δεν θα πρέπει όμως να πέσουμε στην παγίδα τα αποτελέσματα να τα αξιολογήσουμε μόνο με βάση νούμερα. Γιατί τα αποτελέσματα τις δράσεις στον πολιτισμό ε, δεν μπορούν να μετρηθούν μόνο με χρήμα. Είναι σαν να επενδύουμε στο μέλλον. Οπότε αυτό θα πρέπει νομίζω να το υπογραμμίσουμε. Το πώς θα γίνει η αξιολόγηση, η εκτίμηση, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η Χέλγα Τρούπελ έχει το λόγο. Ευχαριστούμε Πέτρα, ευχαριστώ τη Σίλβια και τους άλλους και οδησηγητές. Θα ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση. Όταν ε, συζητάμε το νέο πρόγραμμα για τη Δημιουργική Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε εμείς εδώ και το Συμβούλιο ότι η πολιτιστική πικρομορφία και ο ε, διάλογος μεταξύ διαφόρων πολιτισμών είναι η ουσία της Ευρώπης. Οπότε με τα όσα είπε η Σίλβια. Θα πρέπει αυτό το εργαλείο να συνδυαστεί με άλλες μας πολιτικές. Ο Σίλβια το ξέρει καλύτερα ότι ο πολιτισμός επηρεάζει και βοηθάει την ενδοκατανόηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Silicon Valley είχαμε δει ένα πόστερ που έλεγε «Είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά θέλουμε να μας φέρονται ισότιμα». Ο πολιτισμός οδηγεί προς αυτό. Ναι, δεν είμαστε ομοιογενείς, έχουμε ποικιλομορφία, αλλά από την άλλη μεριά όλοι θέλουμε καλό βιωτικό επίπεδο και δικαιοσύνη. η μάχη με το πολιτιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι πολύ δύσκολη. Ήταν τόσο δύσκολη η διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά την ευελιξία που δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Αν δεν αυξήσουμε τον προπολογισμό μας όμως, όλες μας οι φιλοδοξίες για τα μέσα ε, επικοινω... Ε, επινημέρωσης, για τον πολιτισμό, για την παιδεία κλπ. θα υποσκαφθούν. Θα κινδυνεύσουν. Συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν. Η πολιτισμός μέσα και διατομεακή ενίσχυση είναι η τρεις πυλώνες στους οποίους ε, θα πρέπει να διαρθρώσουμε την ε, γνωμοδότησή μας. Ε, η μουσική είναι πολύ σημαντική. Η μουσική ακουμπάει τις αισθήσει των ανθρώπων, οπότε θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε, να υπογραμμίσουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα για τη μουσική. Και αυτό είναι καλό και για την Ευρώπη και πιο πέρα. Καλό είναι λοιπόν να προσθέσουμε ένα ποσό για τη μουσική. το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε πει, είναι προφανές, είναι φανερή ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα για το θέμα των μικροσχεδίων, μικρό project. Είναι σαφές ότι χρειάζεται συνδυασμό, ισορροπία. κάποιοι συνάλφοι θέλουν πιο μεγάλα project. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε πολλούς καλλιτέχνες, ηθοποιούς, νέους και για να γίνει αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε το πόσο σημαντικά είναι τα μικρο project για την πολιτιστική πλειομορφία στην Ευρώπη. Δεν μου αρέσει η ιδέα του παρατηρητήριου. Πιστεύω θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα όργανα που ήδη υπάρχουν Οπότε οι τροπολογίες μου θα αφορούν τα όσα σας είπα μόλις τώρα. Ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι πάρα πολύ σημαντικός, θα πρέπει να απογραμμιστεί, αλλά να γίνει σαφές ότι αυτό βασίζεται στο κράτος δικαίου. Ε, στην σημερινή πολιτική συγκυρία, κάθε φορά που μιλάμε για κουλτούρα, θα πρέπει να διευκρινίζουμε ότι μιλάμε για δημοκρατικές κουλτούρες και σε κάποια κράτη-μέλη αλλά και εκτός Ευρώπης υπάρχουν τάσεις που απομακρύνονται από αυτή την ιδέα. Εμείς θα πρέπει να το τονίζουμε ότι ο πολιτισμός ενώνει, μιλάμε για διάλογο, αλλά διάλογο μεταξύ δημοκρατικών πολιτισμών και πολιτιστικών παραδόσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αντινόβη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και από στρατηγικής πλευράς γιατί είναι μία από τις λίγες ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους καλλιτέχνες και γενικότερα στον καλλιτεχνικό κόσμο είναι ένας τρόπος να στηριχθούν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ενός τομέα που αντιμετωπίζει πολλά πολλά εμπόδια. Για παράδειγμα, ο ανταγωνισμός εκ μέρους των πολυεθνικών. Υπό το φως όλων αυτών και δεδομένη σημασία του κλάδου αυτού, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα αναφέρονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι τροπολογίες μου έχουν ως στόχο να ευνοηθούν οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες και όλοι όσοι εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο. Καταρχήν πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό. Και το λέω μα. Ένας πρώην, Ιταλό, ε, πρώην Ιταλός πρώην υπουργός έλεγε ότι η κουλτούρα δεν τρώγεται. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι η αύξηση του, η, ο πολιτισμός, η κουλτούρα μπορεί να βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνία και να ευνοήσει ε, την ε, οικονομία. Επίσης, πρέπει να στηρίξουμε τις μικροεπιχειρήσεις. και τις, μικρομεσαίες, και τις μικροεπιχείρησεις και τις μικρομεσαίες. Ε, θα πρέπει να προβλέψουμε ειδικέ ενισχύσεις για όλες τις επιχειρήσεις που προέρχονται από περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ε, όπως οι σεισμοί. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό αυτών που πλήττονται από τέτοιες θεομηνίες. Να τους δείξουμε ότι δεν είναι μόνοι τους, ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να τους βοηθήσουμε αλληλέγγυα Επίσης, είναι σημαντικό να εισάγουμε και κάτι σε σχέση με την προσβασιμότητα, την προσπελασιμότητα των πολιτιστικών αγαθών. Δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις. Αυτό το λέει και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και πολλές διεθνείς συμβάσεις. Θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί η πολιτική μας κληρονομιά και να επενδύσουμε σε νέα φορμάτ και πολυμεσικό περιεχόμενο, multimedia. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσες δυνατότητες έχουμε στα χέρια μας για να δημιουργήσουμε, για παράδειγμα, ένα ευρωπαϊκό Netflix. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Madame. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Βεβαίω και είμαστε υπέρ τη Creative Europe, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα μέσα. Στα θέματα της συμπαραγωγή, ε, της διανομής, ε, της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής, όλα αυτά είναι κρίσιμα. Έχουμε όμως κάποιες αμφιβολίες για την διαφορετικότητα του προγράμματο υπό την κάλυψη τη συνέργεια ή ε, επιχειρησιακής δραστηριότητας διατομεακής έχουμε ε, κάποιες δεσμεύσεις 200 εκατομμύρια ευρώ ε, που κατευθύνονται προς τα μεταναστευτικά ώστε να προεγάγουμε την διαφορετικότητα της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς δηλαδή θεατρικά έργα που να βασίζονται στη ζωή των μεταναστών ή των προσφύγων. Υπάρχουν και, κάποιες, και κάποια βίντεο στο YouTube που κυκλοφορούν σχετικά με αυτά. Ως προς συνεργασία με τις τρίτες χώρες δεν μπορούμε αφενός να λυπόμαστε για την, ε, τις ε, συνεχείς περικοπές του προϋπολογισμού και μετά να ζητούμε όλο και περισσότερα να πετύχει αυτός ο μειωμένος προϋπολογισμός. Έχουμε εδώ κάποιες ε, επιχειρήσεις που υποτίθεται ότι θα υποστηρίζουν τους λιγότερο ανεπτυγμένους, συνόδους στην Τίνισα και στο Κίεβο, με τη ε, συμμετοχή της Αρμενίας, του τα κτλ. Πολύ διασκεδαστικές εκδηλώσεις όλα αυτά, αλλά ε, ε, πρέπει να δούμε τη χρησιμότητά τους στο πλαίσιο των περικομπών προϋπολογισμού που αντιμετωπίζουμε. Εδώ από ό,τι φαίνεται διώχνουμε ή δεχόμαστε την φυγή του Ηνωμένου Βασιλείου και δεχόμαστε με ανοιχτές αγκάλες το κοτσοφοπέδιο. Δεν καταλαβαίνουμε την λογική όλων αυτών των κινήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σκιώδης εισηγήτριά μας, η κυρία Μίχελς, μου ζήτησε να την αντικαταστήσω. Μου, έδωσε γραπτά τις παρατηρήσεις. Με την άδειά σας θα, θα ήθελα να τις διαβάσω. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Σίλβια Κώστα It's okay. Είναι οι παρατηρήσει που μου έδωσε η κυρία Μίχελ. Και τι διαβάζω για να είναι γνωστή η πρώτη μα θέση. Ναι. Ευχαριστή την κυρία Σίλβια Κώστα, η οποία έχει κάνει σημαντικέ προτάσει στο πρόγραμμα Creative Europe. Πέντε παρατηρήσει έχει. Πρώτον, χαιρετίζουμε τον πραγματικό διπλασιασμό του προπολογισμού σε 2,806 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερέ τιμέ και την ποσοστία κατανομή του στι γραμμέ του προγράμματο. Δεύτερον, χαιρετίζουμε την πρόθεση της ελεύθερης δημοσιογραφίας, η οποία περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής με την αιτιολογική σκέψη 12 και το άρθρο 6 γ, καθώς και τις προτάσεις του εισηγητή πάνω σε αυτό. Δυστυχώς αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Τρίτο, χαιρετίζουμε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για, τις, για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Τέταρτο, έχουμε ένα πρόβλημα σε μια διατύπωση, αλλά δεν γνωρίζουμε αν είναι κάτι περισσότερο από ένα γλωσσικό πρόβλημα. Η φράση πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας, όπως προτείνει η Επιτροπή, είναι σημαντική για μας. Ωστόσο, στη γερμανική έκδοση του σχεδίου έκθεσης, έκδοση του σχεδίου έκθεσης, ο όρος πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας αντικαθίσταται συνέχεια με μια τροπολογία από τον εισηγητή, με αποτέλεσμα ο όρος να γίνεται Πολιτιστικέ και δημιουργικέ βιομηχανίε. Αυτό γίνεται σε πολλέ τροπολογίε και σε νέε παραγράφου όπω την τροπολογία 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 αλλά μετά και στα άρθρα. Έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Αν η έννοια του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα έχει αντικατασταθεί με τον όρο πολιτιστικέ και δημιουργικέ βιομηχανίε. Παρακολουθούμε την πρόθεση των πολιτιστικών βιομηχανιών, αλλά ο όρο τομέα είναι ευρύτερο και περιλαμβάνει περισσότερα από ένα είδη οικονομία, ενσωματώνοντα επίση τι δημόσιε υπηρεσίε και την ιδιωτική παραγωγή. Και πέμπτη παρατήρηση, για εμά, το πρόγραμμα Creative Europe πρέπει να δημιουργήσει βιωσιμότητα των υποδομών για ποικίλε πολιτιστικέ λειτουργίε, για ψηφιακή προσβασιμότητα και για τα μη κερδοσκοπικά και δημόσια αρχεία, καθώ και για του ιδιωτικού καλλιτέχνε. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο η έννοια του τομέα είναι πολύ σημαντική για μα. Έρχεται πιο κοντά στη σύμβαση τη UNESCO για το διπλό χαρακτήρα των πολιτιστικών παραγωγών και δεν θα εγκαταλείψουμε αυτή την προσέγγιση. Αν πρόκειται μόνο για ένα γλωσσικό πρόβλημα, θα πρέπει να το λύσουμε. Αν όμω υπάρχει πίσω από τι γλωσσικέ εκδόσει ένα ουσιαστικό ενιολογικό πρόβλημα, πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό και ελπίζουμε ότι θα, μπορέσουμε, θα μπορέσουμε να το βρούμε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δούμε αν όντω είναι θέμα μετάφρασης μόνο. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Όχι, οι, τροπο, τροπολογίες που υπέβαλε η Σίλβια στο σχέδιο, προφανώς στα γερμανικά κάτι άλλο λέει. Μάλλον είναι μεταφραστικό το πρόγραμμα. Το πρόβλημα θα το, θα το ελέγξουμε. Λοιπόν, δεν έχω άλλον που να ζητά το λόγο, οπότε να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, περιμένετε μισό λεπτό γιατί θα έχουμε κι άλλον ομιλητή. Συγγνώμη, έχετε το λόγο. Πολύ γρήγορα, Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να αναφερθώ στο κουσουφοπέδιο, διότι άκουσα στις διακοινοβουλευτικές μας επαφές ε, και σήμερα κάποια δυσάρεστα σχόλια. Ε, μερικοί είμαστε και στην Επιτροπή την διακυλοβουλευτική για τις επαφές με το κοσυφοπαίδιο και είδαμε από την πλευρά τους ε, την πιο θαυμάσια δέσμευση για τα θέματα του πολιτισμού όπου είχαν και μια θαυμάσια έκθεση του Grayson Perry ο οποίος βέβαια είναι Βρετανός καλλιτέχνης, λέει Μιλήτρια. Αλλά νομίζω ότι αν είναι να μιλούμε, να τοποθετούμαστε με, μια, με έναν τρόπο ώστε να αποκλείουμε κάποιες χώρες ε, που αισθάνονται ευρωπαϊκές και που εμείς ή κάποιοι από εμά δεν τις θεωρούν τέτοιες, νομίζω ότι αυτό είναι επικίνδυνο. και μάλιστα ε, η υπεύθυνη του φορέα ε, του πολιτισμού της Πρίστινα είχε διαφύγει από τις σφαγές λεωμιλήτρια στο Μάντσεστα, σε δική μου χώρα. Είναι καλλιτέχνης, είναι ακτιβίστρια, είναι Κοσοβάρα, Βρετανή και Ευρωπαία. Σεράντα Μπογκντοεύσκη, και ε, ελέγξτε την, εδώ μιλούμε για τους γείτονέ μας. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια τοποθέτηση πολύ πιο θερμή απέναντί τους. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα είναι η ώρα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, έχουμε δύο εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της δομής του προγράμματος από δύο γενικές διευθύνσεις από την Γενική Διεύθυνση Air και από την Γενική Διεύθυνση Connect και ξεκινούμε με την κυρία Μπάρμπαρα Γκέσλερ. Έχετε το λόγο. Ε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ και την κυρία Κώστα για την πολύ καλή συνεργασία. Μόνο να το επαναλάβω μπορώ Πραγματικά και εμεί ε, εκτιμούμε πολύ το γεγονός ότι μπορούμε ε, αποτελεσματικά να δουλέψουμε επικοδομητικά για την βελτίωση του προγράμματος. Οπότε, ευχαριστώ και εξ ονόματο της Γενικής μας Διεύθυνση για όλες τις παρατηρήσεις που έκαναν ε, τα μέλη της Επιτροπής σας. τα οποία σίγουρα θα τα δούμε και στην τελική τους εκδοχή την επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για κάποια σημεία τα οποία ήδη ε, προτάθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής. Καταρχάς ευχαριστώ για τη στήριξη για την ε, τομεακή προσέγγιση στον ε, τομέα της, που έχουμε επιλέξει για τον τομέα του πολιτισμού. Σίγουρα αυτό οφείλεται και στο ότι πολλοί από εσάς που είστε και εδώ ή κάποιοι που δεν είναι σήμερα εδώ, όπως ο βουλευτής που έγινε δήμαρχος, ε, είναι σημαντικό αυτό το Music Moves Europe, αυτή την ε, ε, πρωτοβουλία να την υποστηρίξουμε. Πολλοί την έχουν υποστηρίξει και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που την βρίσκεται. Καλή προσέγγιση και η σωστή κατανομή του προπολογισμού δράση θα είναι ένα θέμα που θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε όταν θα ξέρουμε πόσα ακριβώς χρήματα θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά χαίρομαι που εσείς ουσιαστικά συμφωνείτε μαζί μας ότι κάποιοι τομείς θα πρέπει να προωθηθούν ε, λίγο περισσότερο μέσω οριζόντιων ε, project. Όπως είπε και η κυρία Κώστα στην έκθεσή της, θα πρέπει να δούμε και τον τομέα των ε, δημοσιεύσεων, Επίσης να δούμε τι γίνεται με, τον, ε, με το θέατρο και τη, τους ε, καλλιτέχνες, γιατί δεν ε, τους θεωρούμε ως ένα ξεχωριστό κλάδο. Και βεβαίως για, την, ε, για τις παρουσιάσεις, για τους ερμηνευτές, για τους καλλιτέχνες, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πρόγραμμα ίσως πιλωτικό, ώστε μεταξύ των ε, διαφόρων ε, πολιτιστικών βιομηχανιών, δημιουργικών βιομηχανιών να υπάρξει μια ισότητα όπλων και ευκαιριών. Επίσης ευχαριστώ για την στήριξή σας για τον τομέα των διεθνών θεμάτων. Θα δούμε τις ε, προτάσεις για το πώς θα το ονομάσουμε τελικά και ευχαριστώ και όλους τους υπόλοιπους βουλευτές που για τον ε, διακοινοβουλευτικό διάλογο ε, συνειδητοποίησαν ότι αυτό είναι ένα, ένας τομέας που στο τρέχον πρόγραμμα ε, λαμβάνει την προσοχή που του αναλογεί και αυτό δείχνει ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε και τις χώρες της Μεσογείου με συγκεκριμένες στοχευμένες δραστηριότητε και στα Βαλκάνια και για τα ε, χρόνια που έρχονται. Γιατί θεωρούμε ότι για τις ε, σχέσεις γειτονίας της Ευρώπης είναι ιδιαίτερο σημαντικό αυτό. Χαίρομαι δε ιδιαίτερο για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, αύξηση του προπολογισμού. Φυσικά είναι λογικό αυτό. Μιλάμε για μια επένδυση στον πολιτισμό που θα βοηθήσει την Ευρώπη να προχωρήσει. Θέλω να κάνω και δύο σχόλια και αργότερα η Λουσία θα σας κάνει κάποια επιμέρους σχόλια. Στην έκθεση, κυρία Κώστα, προτείνεται να έχουμε ένα παρατηρητήριο. Κάποιοι από τους συναδέλφους σας είπανε ότι δεν υποστηρίζουν την πρόταση αυτή ή τέλο πάντων είναι κάπως σκεπτικοί προς το παρόν. Εμείς μας ενδιαφέρει πολύ να έχουμε σταθερούς και αποτελεσματικούς δείκτες για την αξιολόγηση του προγράμματός μας. Το ίδιο βεβαίως ισχύει σε παρένθεση και για την αξιολόγηση των επιμέρους project. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η ιδιαίτερη ανάγκη του Κοινοβουλίου είναι να έχουμε σωστούς δείκτες, σωστά στοιχεία για να μπορέσουμε να μετρήσουμε αν το πρόγραμμα πάει προς σωστή κατεύθυνση, αν όντως τους στόχους που έχουμε θέσει μπορούμε να τους πετύχουμε. Θα θέλαμε λοιπόν ως προς αυτό να δούμε διαφορετικά μοντέλα για να δούμε πώς μπορούμε όντως να ενισχύσουμε την προσέγγιση. Υπάρχει ας πούμε μια πρόταση του καθηγητού Λουίτζι Σάκο που μας μιλάει για ένα πιλωτικό project ε, ε, που θέλει να ξεκινήσει για την ε, συλλογή δεδομένων μέσω, των, μέσω πληροφορικής με, open, με software open source. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες επαφές που έχουμε με διάφορους οργανισμούς και τα επόμενα χρόνια σίγουρα θα δούμε πώς μπορούμε για τον τομέα του πολιτισμού τέτοιου είδους δεδομένα να τα αυξήσουμε, να τα βελτιώσουμε. Ακόμα και σε περίπτωση που δεν έχουμε τελικά το παρατηρητήριο. βέβαια η Λουσία θα σα κάνει κάποια επιμέρου σχόλια ω προ αυτό για τη δική τη εμπειρία από τον τομέα των οπτικοακουστικών. Ε, σταματώ εδώ για να μιλήσει και η συνάδελφο. Ευχαριστώ. Λουσία, σας ακούμε. Uh, thank you. Thank you very much. Um, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Να ευχαριστήσω και πάλι για την έκθεση, για τα πολύ χρήσιμα σχόλια. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα πρόγραμμα που θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την πρόταση διπλασιασμού του προϋπολογισμού του προγράμματος αυτού. Για τα μέσα επικοινωνίας το έθεσε πολύ εκφραστικά κυρία Κώστα είναι ένα θέμα εξέλιξης. Ε, οικοδομούμε επί προηγουμένων βάσεων, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι προσπαθούμε να καλύψουμε διάφορες αφηγηματικές πτυχές, animation, ντοκιμαντέρ, φιλμ και νέα φορμά, εικονική πραγματικότητα και ούτω καθεξής. Ε, συμφωνούμε ότι είναι στην καρδιά της πρότασης η ανεξάρτητη παραγωγή και δυνομής και είναι κάτι που υποστηρίζουμε απολύτως και για το μέλλον. Για τις τρίτες χώρες θεωρούμε ότι η διεθνής διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά το είχαμε καταστήσει σαφέστερο από ότι στον παρόν κανονισμό ότι οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση της ε, Connecting Europe είναι ο σχετισμός των υποχρεώσεων στην οδηγία οπτικοακουστικών και στην πρόσβαση στις τομεακές διατάξεις της Creating ε, Europe που θεωρούμε ότι είναι μια πολύ χρήσιμη διευκρίνηση για την νέα πρόταση. Επίσης ε, χαιρετίζουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις για τη δημοσιογραφία. Είναι κάτι που είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι χρειαζόμαστε Δηλαδή υποστηρίζουμε, χρειαζόμαστε μάλλον έργα που υποστηρίζουν τον πλουραλισμό και τον αλφαβητισμό των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα πλαίσια των τάσεων fake news που βασιλεύουν, λέγει η ομιλήτρια. Σημεριζόμαστε επίσης τους στόχους ε, του Κοινοβουλίου για την ε, συλλογή ε, στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις πολιτιστικές πολιτικές γενικά και θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να διαματίσει σημαντικό ρόλο εδώ. Θα θέλαμε να ενισχύσουμε την συνεργασία με υφιστάμενες δομέ, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων, που είναι βεβαίω εταίρο και παρέχει πολύ σημαντικά δεδομένα, γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν είχε γίνει μια απόπειρα διεύρυνση της εντολή. Βεβαίω απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν να διατηρηθεί γενικά ω οπτικοακουστικό μέσο φορέα και να μην επεκταθεί σε άλλα πεδία. Επίσης συμφωνούμε μαζί σας ότι η διευκόλυνση ήταν επιτυχής και θα έχουμε περαιτέρω επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες όχι μόνο ή στο πλαίσιο των μικρών και μεσαίων παραθυ... Ε, επιχειρήσεων, με συγχωρείτε, αλλά και του InvestEU. Θεωρούμε πάντως ότι είναι πολύ σωστό και χρήσιμο να δίδεται επιφάνεια σε αυτό το επιτυχές μέσο που είναι η Guarantee Facility, στα πλαίσια της επόμενης ε, ΠΔΠ. Ευχαριστώ. Να δώσουμε και πάλι το λόγο στη Σίλβια. Να ευχαριστήσω λοιπόν για τα σχόλια, και της αιτής ε, που θέλω να δώσω αμέσω. Για την κυρία Ράιαν ε, και εμάς ε, δυσαρεστεί πολύ που για την αποχώρηση του Μπρούνο Βέιντα ξέρουμε ότι θα πάει να κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, είμαι σίγουρο ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί. Τώρα, η διαφήμιση. Το θέμα του παρατηρητηρίου και έτσι απαντώ και σε άλλα σχόλια. Πρέπει να σας πω ότι ως ηγέτρια ήδη στο, στα πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος είχε ανακύψει η αναγκαιότητα σε δημιουργικό καλλιτεχνικό πλαίσιο να μπορούμε να εντοπίζουμε ε, όχι μόνο ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και όλα αυτά να επικαιροποιούσαμε με την έρευνα που υπάρχει σε διεθνές πλαίσιο. Μετά δεν τα κάναμε αυτά γιατί είχαμε πει θα δούμε ε, της κατεξιότητας πράξης. Τώρα μέσα στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι πολύ αυτό. Ε, στο μεταξύ, όλοι οι φορείς θεωρούν τελείως ανεπαρκές το επίπεδο των κριτηρίων αξιολόγηση που χρησιμοποιούνται. Και μιλούμε για τα τρία στοιχεία αξιολόγηση που είναι όλα ποσοτικά. Αυτό δεν είναι δυνατόν υπό το φω τη συζήτηση που είχαμε τον τελευταίο χρόνο για τον διαφορετικό αντίκτυπο των θεμάτων πολιτισμού και για να μην μακρηγορώ. Στο άρθρο 9 και απαντώ στην Σαμπίνε και σε άλλους συναδελφούς, δεν μιλούμε για κάποια καινούργια πραγματικότητα, μιλούμε για την υποστήριξη υφισταμένων πλαισίων. Όπως το πλαίσιο της ερεύνης, της αριστείας της ερεύνης κτλ. Όχι ώστε όλα αυτά να υπάρχονται σε εσωτερικού ερευνητέ, αλλά σε δίκτυο με τα κέντρα ληστεία που έχουμε στην Ευρώπη. Δεν δεν μιλούμε για μια νέα δομή με νέο κόστος, αλλά μια διασύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο. Από εκεί και πέρα μπορούμε να αξιολογήσουμε τους χρόνους και τι διευθετήσεις, αλλά ήθελα να το διαφημίσω. Συμπληρωματικότητα, δεύτερη διευθύνση προσπάθησε να την τοποθετήσω παντού, ιδιαίτερα και στο InvestEU και απαντώ και στην κυρία Τρούπελ. Εγώ ανησυχώ ότι η InvestEU θα μπορούσε να ακυρώσει τροποντινά τις ιδιαιτερότητες που είχαμε θέσει ε, στα πλαίσια του προηγούμενου κανονισμού. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε να επιφέρουμε μια συμπληρωματικότητα των αρχών του InvestEU. Όπως σε αυτό που αναφερθήκατε για τα άλλα προγράμματα, Erasmus, Horizon, ε, κοινωνικό ταμείο, διαθροτικά ταμεία, ψηφιακό. Ε, ε, είναι ένα συνολικότερο πλαίσιο αρκετά δεσμευτικό. Ε, τρίτον, το τμήμα των πολιτιστικών, το θέμα της μικρής κλίμακος έργων, που είπε και η κυρία Τρούπελ και η, η Σαμπίν Φεράιαν δεν μιλούμε για διακριτές διαδικασίες διαγωνισμών, αλλά μιλούμε όταν έχουμε μικρή κλίμακα ή μικρό προγράμματα, έργα, και το δείχνει και η πολύ πρόσφατη εμπειρία μας, να έχουμε μία πρόσθετη συγχρηματοδότηση. Χρηματοδότηση δηλαδή που τα μικρή κλίμακος έργα δεν μπορούν να βρουν στην αγορά. Άλλο ένα στοιχείο. Ζητούμε επίσης μια συγκεκριμένη αφιερωμένη πλατφόρμα για τους ενδιαφερομένους φορείς που ασχολούνται με την πολιστική κληρονομιά για να δώσουμε μια συνέχεια και σε αυτό το διάλογο μεταξύ των ε, μερών. Ήθελα από νωρίτερα να πω ότι εμείς ζητούμε σε κάθε περίπτωση κατέξοδο της συμπράξης γιατί χρειαζόμαστε μια ισορροπία συνομοθεσίας, ως συνομοθέτες δηλαδή. Και άλλη μια απάντηση που άκουσα από πολλού από εσά, το θέμα το τομεακό. Δεν ξέρω αν είναι θέμα γλωσσικό ορολογίας εδώ. Μιλούσα για δημιουργικού και πολιτισμικούς τομεί. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποιήσει εγώ ε, στο ιταλικό κείμενο. Τώρα δεν ξέρω τι, μεταφέρθηκε και άκουσα για τα τομεακά. Ε, το νέο ζήτημα του υποστήριξης της ποιοτική δημοσιογραφίας του κριτικού πνεύματος. Όλα αυτά τα, τα ενσωματώσαμε για να καλύψουμε και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ σημαντική η συμπερίληψη ε, της μνήας στις γυναίκες, της θηλυκής οπτικής γονέας, ε, τα φύλλα. Και επίσης σημαντικό, και νομίζω ότι απάντησα στο θέμα για την σχετισμό με την διεθνή διάσταση, Νομίζω ότι έχουμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη μας τη νέα διεθνή καλλιτεχνική δημιουργική στρατηγική και αυτή την προσθήκη του Μούντους θα μας προσέφερε μια διάδραση με τα όσα συμβαίνουν σε πολιτιστικό πλαίσιο διεθνώς. Είχαμε επικαλεστεί και διμερείς συμφωνίες των χωρών της Ευρώπης με τρίτες χώρες γιατί είναι πολύ λίγες αυτές που συμμετέχουν επί τη βάση ιδίων πόρων και να απαντήσω και στους συναδέλφους που αναφέρθηκαν. Υπογραμμίσαμε πάρα πολύ την σημασία συνολικά του πολιτισμού, της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας καλλιτεχνικής έκφρασης δηλαδή και δημιουργίας Και το κάναμε όπως το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά προσθέσαμε τα τις οδηγίες επί των οπτικοακουστικών, γιατί είναι άλλο ένα μέσο που μπορεί να μας βοηθήσει. Και επομένως υπογραμμίσαμε, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο το νέο νομοθετικό ε, πλαίσιο, στο οποίο, μάλλον, στο οποίο θα πρέπει να υπάρχονται ή συμμετέχονται στο πρόγραμμα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους. Περιμένω με ενδιαφέρον τις ε, τροπολογίες. Θα τις διαβάσουμε με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ τις, ε, τους εκπροσώπους των δύο Γενικών Διευθύνσεων της Κομισιόν και πραγματικά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε ε, να έχουμε μια δημιουργικότατη δουλειά. Ευχαριστώ βεβαίω και την Γραμματεία για την υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Σίλβια. Ε, προθεσμία για τις ε, τροπολογίες 29 Νοεμβρίου στις 3 το απόγευμα και Εύχομαι στη Σίλβια και στους σκιώδες ηγητές της καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία στην περαιτέρω εκπόνηση του προγράμματος. Και όταν ε, θα έχουμε και τον ε, προποδορισμό θα δούμε πώς θα παίξει και αυτό στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, παρουσίαση της έκθεσης Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή και τα επόμενα βήματα. Μιλούμε για την υποβολή λοιπόν της έκθεσης της Κομισιόν για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊάννα και του τρόπου με τον οποίο θα προχωρήσουμε από εδώ και μπρο επί τη βάση μιας ανεξάρτητης μελέτης. Η μελέτη αυτή μας δίνει ε, συγκεκριμένα στοιχεία και συμπληρωματικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της Ευρωπαϊάννα και περιλαμβάνει και κάποια βήματα ε, καθοδήγησης για την πελωτική εξέλιξη του προγράμματος. Ξέρετε ότι η Επιτροπή μας ε, την εξέλιξη τη Europeana από την αρχή της δημιουργίας της εδώ και μια δεκαετία το υποστηρίζει εντατικά και την παρακολουθεί προσεκτικά. Η παρουσίαση αυτή λοιπόν τη έκθεση για μα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα ήθελα να χαιρετήσω, να καλωσορίσω την κυρία Ρεάνα Σβίνιγκα Λαντάκ, η οποία είναι η προϊσταμένη της Μονάδας Δραστικών Τεχνολογιών Ψηφιακού Πολιτισμού και Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Connect, η οποία θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης. Κυρία Σβίνιγκα, Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που είστε εδώ. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ονομάζομαι Σφίνιγκερ Λάντακ και είμαι τη συνάδελφό μου για να σας παρουσιάσουμε την αξιολόγηση της Κομισιόν για την ε, Ευρωπαϊκή. Μιλάμε για τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτιστική ποικιλομορφία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία συζητούμε συνεχώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την ψηφοφορία στην έκθεση για την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Ε, έχω και την ψηφιακή εκπαίδευση στην αρμοδιότητά μου, ιδιαίτερα την, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων σε μια εποχή που η ψηφιακή τεχνολογία καλπάζει. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ότι μας ε, στηρίξατε σε θέματα συνδεσιμότητας, ότι τα σχολεία θα πρέπει να ε, είναι συνδέσιμα και να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ κλπ. Παρουσιάζουμε αυτή την έκθεση στο Κοινοβούλιο τη μέρα ακριβώς που κλείνει 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή. Έξι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων πριν από 10 χρόνια έστειλαν μια επιστολή με την οποία δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή. Είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα που δίνει πρόσβαση σε ψηφιακή πολιτική κληρονομιά με πάνω από 3.700 700 φορείς που συμμετέχουν, αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, συλλογές κλπ. κλπ. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ζωντανό δίκτυο επαγγελματιών και ένα οικοσύστημα φορέων και ατόμων που συνεισφέρουν. Εντάσσεται στην, στο πρόγραμμα Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη, θα σας μιλήσω τόσο περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή η αξιολόγηση λοιπόν είναι πολύ ε, επίκαιρη. Βέβαια, προφανώς το Συμβούλιο μας έχει ζητήσει να εξετάσουμε το πώς, ε, τι επιδόσεις έχει η Ευρωπαϊκή αν υφίσταται ένα μηχανισμό βιώσιμη χρηματοδότηση και ποιε είναι οι συστάσει για το μέλλον, ενώ ταυτόχρονα στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κουλτούρα ήδη ανακοινώσαμε αυτή την εκθεσή μας και τέλος είναι επίκαιρη διότι όταν εξετάζουμε το ε, σε μια εποχή που εξετάζουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την νέα περίοδο είναι καιρός και ευκαιρία να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον με το πρόγραμμα αυτό. Οπότε μπορούμε να κοιτάξουμε τι έγινε στο παρελθόν, ποιε ήταν οι αδυναμίε και τι θέλουμε να γίνει στο μέλλον. Το πεδίο της αξιολόγησης ε, καλύπτει την έννοια και την αξία της ευρωπαϊκής ως ευρωπαϊκό πολιτιστικό project και project ψηφιακής κρινοτομίας και τα δύο δηλαδή. Ταυτόχρονα εξετάζουμε την επάρκεια και την βιωσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή. Η αξιολόγηση έγινε με σεβασμό των ε, πέντε υποχρεωτικών ε, κριτηρίων για την ε, βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης μας στήριξε ε, ένας, ε, μια ανεξάρτητη έκθεση η οποία έγινε εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πέντε ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες από που κάθε ένας ε, αντιπροσωπεύει μια διαφορετική πτυχή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Επίσης, είχαμε διάφορες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες συνεισέφεραν σε αυτήν την αξιολόγηση. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει προφανώς το σώμα της έκθεσης που συνοψίζει τα πορίσματα και δίνει μια ιδέα για το ποιο είναι το όρμα για το μέλλον και ένα έγγραφο εργασία με περισσότερα στοιχεία. Ταυτόχρονα διανοηγήσαμε και μια διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση στο ίντερνετ. Πήραμε πολλές απαντήσεις πάρα πολύ feedback και πολύ πάθος. Χρειάστηκε βέβαια να φιλτράρουμε το, το πάθος, <laughs> αλλά οι συνεισφορές ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες. Και τι μας λένε όλα αυτά. Υπάρχουν, έχει και ε, μεγάλα προτερήματα και αδυναμίε η Ευρωπαϊκή. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή είναι η μοναδική πανευρωπαϊκή πλατφόρμα και μοναδική στο είδος της στην Ευρώπη. Αποτελεί την μεγαλύτερη ψηφιακή συλλογή από τα 28 κράτη-μέλη, πάνω από 60 εκατομμύρια ε, αντικείμενα επίσης εμπνέει το αίσθημα της κοινή ιστορίας, του κοινού παρελθόντος, ε, Έχουμε εκστρατεία για τις μεταναστεύσεις, σε, μερικές, σε μερικούς μήνες θα έχουμε μια εκστρατεία για τις γυναίκες, για την επιστήμη κλπ έχουν συμμετάσχει πάρα πολλοί φορείς και πάρα πολλοί πολίτες. Επίσης μας οδήγησε στο να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές, τις καλύτερες λύσεις και τις καλύτερες προδιαγραφές και γίνεται μια ε, de facto τυποποίηση της κληρονομιάς μας. με δηλώσει, για παράδειγμα, διεθνείς δηλώσεις ε, δικαιωμάτων κλπ. Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και αργότερα. Η Ευρωπαϊκή επίσης δημιούργησε ένα ολόκληρο δίκτυο ε, επαγγελματιών και ατόμων και φορέων που συνεισφέρουν στο δίκτυο και επίσης ε, συμπληρώνει τις εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών και υλοποιεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τώρα υπάρχουν κάποιες προκλήσεις Προσπαθήσαμε να είμαστε δίκαιοι. Θέλουμε να καταλάβουμε ποια είναι τα σύνολα αλλά και ποια είναι τα πλήν, ποιε είναι οι αδυναμίε τη Ευρωπαϊκή. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε την Ευρωπαϊκή στο επόμενο πολιτιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει να ξέρουμε ποιε είναι οι προκλήσει που θα αντιμετωπίσει. Και είναι αρκετέ. Πρώτον, ότι το κοινό τη Ευρωπαϊκή είναι πάρα πολύ πλατή. Χρειάζεται να εστιάσουμε περισσότερο τους πραγματικά εμπλεκόμενους με την πολιτική κληρονομιά. Δεύτερον, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία και μεταδεδομένα, αλλά υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ό,τι αφορά την ποιότητα αυτών. Γιατί μέχρι τώρα δώσαμε πολύ βάρος στην ποσότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, στον πλούτο του δεδομένου και του περιεχομένου και των μεταδεδομένων. Κατόπιν η ευρεσιμότητα του υλικού. Είναι πολύ το υλικό και γι' αυτό λόγο δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις αυτό που θέλεις. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, μάλλον χρειάζεται να κάνουμε ε, στο μέλλον πολλές ε, προσπάθειες έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις μηχανές αναζήτησης, να ε, προετοιμάσουμε εργαλεία που θα επιτρέπουν ευκολότερη πρόσβαση και βέβαια πολυγλωσία. Γιατί πολύ συχνά σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχουν οι πόροι για να γίνει μια, ε, ένα localization αυτού του εργαλείου, μια προσαρμογή στην εθνική γλώσσα. Υπάρχει επίσης άλλο ένα, μια πρόκληση ό,τι αφορά το πώς εντάσσουμε τις προβλήσεις που μας έρχονται, ε, καθώς επίσης και την προώθηση της Ευρωπαϊκής στο κοινό το οποίο κοινό δεν είναι πάντοτε ενημερωμένο για την ύπαρξή τη. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία θα εργαστούμε τα επόμενα χρόνια. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας λοιπόν για την Ευρωπαϊκή στο επόμενο πολιετές μεσονομικό πλαίσιο. Έχουμε υπογραμμίσει εδώ τους άξονες στους οποίους θα διαρθρώσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Καταρχήν, Θέλουμε η Ευρωπαϊκή να υπηρετεί τους βασικούς εμπλεκόμενους σε θέματα ψηφιακής πολιτιστικής χρονομιάς. Να στηρίξει την ψηφιακή τους μεταμόρφωση, μετασηματισμό και θα είναι το βασικό εργαλείο για κάτι τέτοιο. Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσουμε την τεχνική πλατφόρμα βελτιώνοντας κάποια τεχνικά στοιχεία όπως η ευρεσιμότητα, η πολυγλωσία, ε, η ένταξη καινούριων πληροφοριών και δεδομένων. Επίσης θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην διαθεσιμότητα του περιεχομένου. Το περιεχόμενο δημιουργείται και από φορείς που ασχολούνται με την πολύ Έχουμε πάρα πολλά τέτοια δεδομένα. Θα πρέπει όμως να, χρησιμο... να δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία σε αυτούς τους φορείς έτσι ώστε να δημιουργούν πραγματικά ελκυστικό περιεχόμενο έτσι ώστε να, ε, να εμπνέει τους χρήστες. Μετά, χρειάζεται να κάνουμε τυποποίηση, να διαδώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, κοινέ λύσεις σε κοινά προβλήματα. Πολύ συχνά οι φορείς δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι ευκαιρίες που τους δίνει η ψηφιακή εποχή. Οπότε η Ευρωπαϊκή θα επανεστιάσει στο να εξυπηρετεί τους φορείς που εμπλέκονται στην πολιτιστική κληρονομιά, την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την Ευρωπαϊκή μέσω του προγράμματος Φιακής Ευρώπης. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας. Σκοπεύουμε να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή επίσης μέσω ενός δικτύου κέντρων ε, αριστείας ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που γνωρίζουν ε, πολύ περισσότερα από κάποιου άλλου ενδεχομένω για την ψηφιοποίηση τη πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, συμπληρωματικά, χρηματοδότηση από, τον, από το ορίζον Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της πρωτοβουλίας αυτής, ε, το μόνο που θα σας πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίξει ε, βασικό συντονιστικό ρόλο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πλήρη η παρουσίασή σας. Μας ε, έδωσε διάφορα στοιχεία, προτάσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε για το μέλλον, πού πρέπει να βελτιώσουμε, πού πρέπει να επικεντρωθούμε όχι τόσο πολύ στα ποσοτικά χαρακτηριστικά, αλλά στα ποιοτικά των δεδομένων, το θέμα της προσβασιμότητας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλες τις λεπτομέρειες που μας δώσατε και ξεκινούμε τη συζήτηση με την Σαμπίνε Φερχάγεν. Ευχαριστώ. Και εκ μέρους του ΕΛΚ ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή όλων των στοιχείων. Μας μιλήσατε και για, τα, για τις προκλήσεις, ε, για εμείς ως Επιτροπή πολιτισμού πάντα θεωρούσαμε ότι ο European είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Βλέπω αυτά που αναφέρατε στα πλαίσια της, ε, των προκλήσεων για την έλλειψη ευαισθητοποίησης. Αναρωτιέμαι, εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί η Europeana, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να την προωθήσουμε στα ε, ιδρύματα, στα σχολεία, γιατί σε αυτά ε, αποτείνεται. Είναι ένα αρκετά αξιόλογο εργαλείο αλλά αν ρωτήσει κανένα στα σχολεία ποιο ξέρει τη Γεωροπεάνα, ούτε οι καθηγητέ ε, καλλιτεχνικών δεν τη γνωρίζουν. Οπότε έχετε κάποιε συγκεκριμένε ιδέε για το πώ μπορεί αυτό να αλλάξει. Και επίση, ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί βλέπουμε διάφορα project κτλ. να τα προωθήσουμε, να τα χρηματοδοτήσουμε, αλλά δεν φτάνουν στου πολίτε. Τελικά είναι δώρον άδωρον, γιατί πραγματικά η Γεωροπεάνα είναι πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Δεύτερο ερώτημα τι γίνεται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για τα θέματα της χρηματοδότησης. Θα μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε την χρηματοδότηση για την δομή. Υπάρχουν προβλήματα με τη χρηματοδότηση. Τι γίνεται. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ Ζαμπίνα. Χέλγα. Ευχαριστώ. Και από τη δική μου την ε, πλευρά πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. και τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊάνα, Συμφωνώ με τα, με τα ερωτήματα της ε, Σαμπίνη, γιατί τώρα έχουμε τα δέκατα γενέθλια της Ευρωπαϊάνα και το ερώτημα που μου έρχεται πρώτα στο μυαλό είναι ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη διαφήμισης, γνώσης, γιατί δεν το ξέρουν οι πολίτες. Ξέρω ότι είναι δύσκολη βέβαια η κατάσταση ό,τι αφορά την, ε, τον ανταγωνισμό με ιδιωτικού παίχτε τη κακέρα, αλλά έχουμε πρωτοβουλίε τέτοιου είδου και τώρα έχει πάψει να είναι με απλή πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή, αλλά καλό είναι να τις προωθούμε τέτοιου είδους ε, ε, πρωτοβουλίες. Οπότε θα ήξερα, θα ήθελα να μου πείτε γιατί δεν υπάρχει η γνώση και πώς μπορεί να αποκτηθεί. Ε, ποιότητα των δεδομένων, προσβασιμότητα, πάντα είναι σημαντικά θέματα αυτά. Και κάτι ενδιαφέρον για μένα, είπατε ότι υπάρχει, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν αρκετά ε, επεξεργασμένα φίλτρα. εγώ ε, ήμουνα σε μία επίσκεψη ε, με παιδιά γυμνασίου ε, και τους ενδιαφέραν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τα φίλτρα. Τώρα μιλάτε για μια πολύ υψηλής ε, ποιότητας, ένα υψηλής ποιότητας φιλτράρισμα, για να μπορεί κανείς δηλαδή να βρει αυτό που ψάχνει, κυρίως ό,τι αφορά τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ίσως ακριβώς επειδή είναι κομμάτι του αγώνα που γίνεται για την πολιτιστική κληρονομιά, θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις μεγάλες πλατφόρμες. Εσείς τι κάνετε για να επενδύσετε σε τέτοιου είδους φιλτράρισμα, ποια είναι αυτά τα φίλτρα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε και πώς τα δημοσιεύετε, πώς σου δημοσιεύετε την ανάγκη να υπάρξουν αυτά τα φίλτρα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Χέλγα. Σίλβια Κώστα. Πρόεδρε, εμεί είμαστε ενθουσιώδει οπαδοί τη Ευρωπαϊκή αλλά κάπω απογοητευμένοι λόγω της, ε, του μεγάλου δυναμικού και του μπλοκαρίσματο κάπως τα τελευταία χρόνια. Όλοι αυτοί που παρακολουθούν το Ευρωπαϊάν ε, μας διηγούνται όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που γίνονται, αλλά υπάρχει μια, ένα κενό που να καλύψουμε, να πληρώσουμε. Νομίζω ότι πολύ σωστά αν να προσανατολίζεται μέσω της αρχής επαφής με κάποιους συνομιλητές. Εσείς τώρα εστιάζεστε στην πολιτιστική κληρονομιά και στις κοινότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και υπό τη Σύμβαση Φάρο, απλώς για να καταλάβουμε καλύτερα. Τώρα, έχουμε και αυτό το δίκτυο διαβούλευσης αλλά στο Ευρωπαϊάννα υπάρχουν και κάποιες διεπαφές ε, εδαφικές, περιφερειακές. Θα μπορούσε δηλαδή να φανταστεί κανείς ε, και κάποιους άλλους ε, φορείς που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε αυτό το δίκτυο, σε αυτό το κύκλωμα, στην μεγάλη οικογένεια Ευρωπαϊάννα. Επόμενες εδαφικές επαφές πρώτον. Δεύτερον, στο επόμενο πι ε, θα είμαστε Digital EU και ε, Horizon. Ε, έχουμε συγκεκριμένες προβλέψεις για τα εκπαιδευτικά, γιατί στα του Cultural Heritage δεν συμπεριλαμβάνονται ακαδημαϊκά ιδρύματα, πανεστήμια. Και τέλος, για τη διαβούλευση, αυτοί που στρέφονται σε εσά, οι φορείς, αυτοί οι 300 όσοι και να είναι, έχετε προχωρήσει σε μια ανάλυση μεταξύ αυτών μια ιεράρχηση ποιοι είναι καλύτεροι γνώστες, ποιοι λιγότερο, ποιο παρακολουθεί, ποιος την τα πράγματα εξ αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σφίνγκα, έχετε το λόγο να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. So, to, to, uh, on the question... Ναι, Πρόεδρε. Για την η ερώτηση του Ευρωπαϊκού και την ενσωμάτωση στη σχολεία εξαρτάται από τις χώρες. Στη Γαλλία π.χ. έχουν συνεργαστεί στενά και προβλέπεται ως πηγή για το σχολικό υλικό, αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν έχουμε ένα ελκυστικό υλικό, ε, είναι δύσκολο να συμμετάσχουν δηλαδή και οι μαθητές να έχουμε το ενδιαφέρον τους. Είναι λίγο παγίδα. Και βεβαίως και κάνουμε την, ε, την διασύνδεση, τη γέφυρα ε, μεταξύ των πολιτιστικών και των εκπαιδευτικών. Για τη χρηματοδότηση. Μέχρι τώρα χρηματοδοτούσαμε το Ευρωπαϊάννα ε, υπό δύο διαφορετικά πλαίσια. Καταρχάς χορηγίες αυτό δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα συγχρηματοδότησης για τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούσαν να σεβαστούν, αν θέλετε, το, τη, δική τους, το δικό τους μερίδιο συγχρηματοδότησης. Πέρυσι το αλλάξαμε αυτό σε προμήθεια γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Έχουμε το, σκοπό, την πρόθεση να συνεχίσουμε με, μια, με ένα ανάμεικτο σχήμα προμήθειας και χορηγία για να μην επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε στο επόμενο πι Δηλαδή να έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας αν θέλετε για τη χρηματοδότηση. Τώρα η σύμβαση που έχουμε είναι προμήθεια για δύο έτη που μπορεί να ανανεωθεί για άλλα δύο. Για το, την ερώτηση της κυρίας Τρούπελ, τι ευθύνεται στην έλλειψη ευαισθητοποίησης. Είναι τόσοι πολλοί παράγοντες που τι να σας πω είναι πάρα πολύ διαφορετική η κατάσταση, εξαρτάται από τη χώρα τη συγκεκριμένη. Σε μερικές χώρες είναι γνωστό, σε άλλες δεν είναι. Το να σας πω γιατί είναι αρκετά δύσκολο. Ίσως και γιατί το έργο της Ευρωπαίαννα εστιάστηκε στην γεφύρωση των ψηφιακών κενών μεταξύ άλλων και ίσως κάποια ενδιάμεσα τμήματα χάθηκαν στον δρόμο, αλλά γνωρίζουμε ότι στις εκστρατείες που έγιναν υπήρξαν πολύ επιτυχείς. Σε, ένα, σε, σε, θεματικές τόσο βαριές, για να το πούμε έτσι, όπως αυτή του Πρώτου Παγκοσμίου, 14-18. Δηλαδή, περισσότερο υλικό που θα μπορούσε να ε, ενισχύσει αυτή την, ε, την αίσθηση της ε, κοινή ταυτότητας για την έλλειψη επαρκών φίλτρων. Σε πολλές θητιακές πύλες με ευρύ περιεχόμενο και συγκεκριμένα για τα πολιτικά θα έπρεπε κανείς να μπορεί να φιλτράρει τα αποτελέσματα. Αν κανείς όμως αναζητά, ψάχνει συγκεκριμένα ντανταϊστές ή ιμπρεσιονιστές, δηλαδή πρέπει κανείς να διαφημίζει τι ακριβώς αναζητεί. Δηλαδή βασικά, βασικοί μηχανισμοί φιλτραρίσματος που θα περιμέναμε σε οποιαδήποτε ψηφιακή πλατφόρμα στο Ευρωπαϊκό να δίνει ακόμα εκεί. Και θα θέλαμε να είναι. Και επίσης η κάλυψη του περιεχομένου είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει περιεχόμενο που επιτρέπει στους επισκέπτες να το διατρέξουν για να ανακαλύψουν τι, περισσότερο υπάρχει. Αυτό είναι συνολικά ε, ένα ζήτημα για το ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά περιεχόμενα και ιδιαίτερα για τα του πολιτισμού. Για την κυρία Κώστα τα, της χρηματοδότησης. Στα πολιτιστικά έχουμε μια συνολική προσέγγιση που είναι αφενός η χρηματοδότηση μέσω του Digital Europe ώστε να ενισχύσουμε τα παρεχόμενα της λειτουργικότητες που θα συμπληρωθεί από το κέντρο δεξιοτήτων. Γιατί θα εξαρτηθεί από, τις, από τεχνολογικό δυναμικό των φορέων των πολιτικών. Αν θέλει κανείς να ψηφιοποιήσει, να κάνει μια μοντέλα, ε, ένα μοντέλο με ε, ε, τρισδιάστατο, μπορεί να πάει σε ένα τέτοιο κέντρο αριστείας, δεξιότητος και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικότερες προκλήσεις έρευνας που θα γίνουν υπό το Horizon. Για την κοινότητα, η κοινότητα νομίζω που έχουμε οικοδομήσει είναι 3.700, σχεδόν 4.000 δηλαδή επαγγελματικοί φορείς που έχουν ήδη δεσμευθεί. Βεβαίως και γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε μια κρίσιμη μάζα για να φτάσουμε στο επίπεδο το τοπικό, το περιφερειακό κτλ. Εμείς έχουμε φορείς από όλα τα 28 κράτη-μέλη, αλλά θέλω να εξασφαλίσουμε ότι κάθε φορέας, ακόμα και πιο μικρός, μπορεί να συμμετάσχει. Γιατί μιλούμε και για την δημοκρατική προσβασιμότητα στην πολιτική κληρονομιά. Για τους φορείς, αλλά και για τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις λοιπόν που ακόμα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άρα πολλή δουλειά έχετε μπροστά σας. Να είστε πάντως σίγουροι ότι η ε, Επιτροπή Πολιτισμού θα είναι στο πλευρό σας. Σίγουρα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, θα παρακολουθούμε αν έχετε προχωρήσει, τι γίνεται με την ευρεσιμότητα τον, ε, του υλικού κτλ. και επίση τι γίνεται σε σχέση με την ε, διαφήμιση τη Europeana και πόσο το χρησιμοποιούν, πόσο ξέρουν το πόρταλ αυτό. Είναι και αυτό ένα σημαντικό σημείο, γιατί το πόρταλ τη Europeana είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν πολύ καλέ πρωτοβουλίε. Σα ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα και μα το παρουσιάσατε. Μα δείξατε σε ποια κατεύθυνση θέλετε να κινηθείτε. Και καλή επιτυχία με την δουλειά που έχετε να κάνετε. Ε, στο μέλλον ε, να είστε σίγουροι ότι η Επιτροπή Πολιτισμού θα είναι δίπλα σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, άρα τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη. Στα διάφορα εγώ δεν έχω τίποτα. Οπότε η επόμενη συνεδρίαση είναι την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα και θα ξεκινήσουμε με την συνεδρίαση των συντονιστών, οι οποίοι γίνονται, συνεδριάζουν και των θυρών, οπότε παρακαλώ όσοι δεν πρέπει να είστε εδώ, να αποχωρήσετε και να κάνουμε ένα μικρό πεντάλεπτο διάλειμμα για να μπορέσουμε να πάρουμε όλοι τις θέσεις μας.